θέμα τη ε, τροποποίηση τη μεστή διατάξεω. Για τη Δευτέρα δεν υπάρχει καμία αίτηση για τροποποίηση. Τώρα, για την ε, Τρίτη, η ομάδα των Πρασίνων ζήτησε Η ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν αναφορικά με την οικονομική κρίση να συμπεριληφθεί στο σχέδιο μεσίας διατάξεως για αύριο στις 15.00. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της ομάδα των Πρασίνων να μα αιτιολογήσει το αίτημα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε που δίνετε το λόγο για το θέμα αυτό. Θεωρώ το προσπαθήσαμε να το συζητήσουμε και μεταξύ των Πρόεδρων των ε, ομάδων ότι το Κοινοβούλιο μετά αυτό το λυπηρό από το Κυριακό των Βρυξελών δεν μπορεί να φύγει από τη συζήτηση για την επίλυση της κρίσης και δεν θα πρέπει να περιμένουμε την πέμπτη να ενημερωθούμε ή μπορεί και όχι για την κατάσταση. Όχι, θα πρέπει να παρέμβουμε κατεπηγόντως. Εγώ έμεινα μάλιστα όλο το Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες και προσπάθησα να ακολουθήσω τις όλες τις αποφάσεις σε όλες τις φάσεις. Μου κάνει λοιπόν πολύ εντύπωση που μία σύνοδος η οποία μετά από 14 μέρες αναβολή ε, λαμβάνει η χώρα και δεν μπόρεσε να πάρει βασικές αποφάσεις. Όσο πιο έντονη είναι η κρίση, τόσο πιο άσχημα εξελίσσεται η ικανότητα συμφωνίας. Όσο πιο βαθιά ε, αναλύεται η κρίση, τόσο και πιο βαθύ είναι το πολιτικό ρήγμα, η πολιτική κρίση μεταξύ των αρχηγών κυβερνήσεων και κρατών στη Σύνοδο. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφής και ξεκάθαρη και νομίζω ότι ενώπιον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό να εκπροσωπήσουμε και να εξηγήσουμε διαρκώς αυτή την ε, ε, θέση, διακόπτει ο Πρόεδρος. Είναι διαφορετική λοιπόν, συνεχίζει η κυρία Χάρμς. Ε, γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι αύριο στην ε, συζήτηση αυτή θα πρέπει να κάνουμε μια δήλωση πριν από τη Σύνοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρόεδρος Σούλτς. Έχετε το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο να μην μάθουμε την Πέμπτη το τι έγινε, γιατί θα τα μάθουμε τα πράγματα αυτά την Πέμπτη όταν θα έχει τελειώσει η Σύνοδος, αλλά να ξεκαθαρίσουμε την θέση του Κοινοβουλίου ως προς την διαδικασία. Θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε χρόνο ε, συνεδριάζοντας μεταξύ των ομάδων για να αποστείλουμε από το Κοινοβούλιο ένα σαφές και ηχηρό μήνυμα προς το Συμβούλιο. Αυτό θα το υποστηρίζει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. E, Ευχαριστώ. Το έτοιμά σα είναι σαφέ. Ε, το διατυπώσατε ξεκάθαρα. Θα πρόκειται για μια δήλωση ε, των πολιτικών ομάδων και φυσικά δήλωση του Συμβουλίου και τη Κομισιόν για να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν άλλοι που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Κατά, κατά ε, τη αίτηση Όχι τότε υποβάλλω προς ψήφιση το αίτημα. Ποιο είναι υπέρ της πρότασης των πρασίνων. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Το αίτημα έγινε δεκτό. Θα τροποποιήσουμε καταλήλως ε, την αυριανή μέσα διάταξη. Αύριο το απόγευμα λοιπόν στις 15.00 θα συμπεριληφθεί το ζήτημα που μόλις ε, ψηφίσαμε. Η συζήτηση θα διαρκέσει περίπου 45 λεπτά και τα υπόλοιπα σημεία, όπως καταλαβαίνετε, θα καθυστερήσουν κατά τρία τέταρτα. Δεν πρόκειται για μια σημαντική χρονικά τροποποίηση, αλλά φροντίσουμε να κατανείμουμε τον χρόνο μας ε, καταλήλως αύριο το απόγευμα και αύριο το βράδυ. Λοιπόν, θα συμπεριλάβουμε αυτό το σημείο στην αυριανή μέσα διάταξη. Προκειμένου για την Τετάρτη και την Πέμπτη δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα τροποποίηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι εγκρίνεται η μέσα διάταξη και μπορούμε να περάσουμε το πρώτο σημείο αυτή. Πρόκειται για την έκθεση Άνταμ Κόσα, κινητικότητα και ένταξη ατόμων με αναπηρίες. Να περιμένουμε δύο-τρία λεπτά πριν να ξεκινήσετε την ομιλία σας, αγαπητέ φίλε, γιατί... You say no. You say no. You say no. Two minutes, please. Δύο λεπτά, δύο λεπτά παρακαλώ. Because our colleagues... Επειδή οι συνάδελφοι φεύγουν από την αίθουσα, δύο λεπτά λοιπόν διάλειμμα. Sorry. Yeah, yeah. Um, um, madam, uh, madam. Uh, η κυρία Λούλινγκ, πρόεδρε, πρόκειται για την ημερήσια διάταξη της Τρίτης. Στην ημερήσια διάταξη αναφέρεται μια προφορική ερώτηση σχετικά με την οδηγία αναφορικά με την μητρότητα. Εγώ εκπλήσωμαι διότι εγκρίναμε την έκθεσή μας σε πρώτη ανάγνωση Βρισκόμαστε στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Καρδιάρκεια της διαδικασίας συναπόφασης δεν υποβάλλουμε στο Συμβούλιο ερωτήσεις ε, για θέματα που άπτονται των παραχωρήσεων που είναι επί της εκθέσεως. Θεωρώ ότι αυτή η ερώτηση δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στη μέση διάταξη. Διαφορετικά δείχνουμε στο Συμβούλιο ότι δεν καταλάβαμε τίποτα από την διαδικασία συναπόφασης και την ε, ε, συνθήκη Λισαβόνα. Ευχαριστώ κυρία Λούλινγκ, ευχαριστώ για, την, για το σχόλιο σας. Θα ελέγξουμε, θα επαληθεύσουμε το σημείο αυτό. Πρόκειται